Συνεχίζουμε λοιπόν τη σύνοδο. Οι αρμόδιες αρχές της Λετωνίας είπαν ότι εξελέγει η κυρία Λιεπίνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντικαθιστώντας τον κύριο Ντομπρόφσκι. και αυτό από τις 19 Μαρτίου 2009 ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού. Εφόσον δεν έχει γίνει επαλήθευση των διαπιστευτηρίων του και δεν έχουν ξεχαστεί τα έγγραφά της μάλλον, κυρία Λιεπίνα θα είναι στο ε, Κοινοβούλιο, θα απολαμβάνει το δικαιωμάτων τη όρου φορή του Κοινοβουλίου. Από τη στιγμή που εκ των προτέρων θα κάνει δήλωση ότι δεν έχει ασύμβατα καθήκοντα με αυτά του Ευρωβουλευτού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Μενήσια διάταξη έχει την προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα ε, για του φορτιστέ ε, κινητών.